Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας, εκεί ακριβώς όπου ε, σταματήσαμε, πριν από το μεσημερινό διάλειμμα δηλαδή. Πρέπει να μιλήσουμε τώρα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και δίνω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή Κονζάλε Πόνς, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του όσον αφορά πάντα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην περιφέρεια Καστίγια Ιλέων της Ισπανίας. Μιλάμε για 700.000 ευρώ. Κινητοποίηση του Ταμείου για το ποσό αυτό. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 η Ισπανία ζήτησε την αρρωχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για να μπορέσουν οι 587 εργαζόμενοι που έχασαν την εργασία τους από τα τέλη 2012 μέχρι το 2013 να βοηθηθούν από πλευράς του τομέα ξύλου και φελού στην Καστίγια Ηλεών. Είναι υποχρεωτικό να ευχαριστήσουμε για τη διαδικασία και εξέταση της αρρωγής αυτής τον ρόλο που διαδραμάτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μέλη αυτής της, ε, της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τουλάχιστον από πέντε κομματικές ομάδες καθώς επίσης ε, και για το Δήμο και τις ε, εργατικές ενώσεις της περιοχής Καστήλης και Λεών. Για το αίτημα αυτό ολοκληρώθηκαν στις 22 Ιουλίου 2014 με συμπέρασμα ότι συμπληρώνονται οι όροι για να κινητοποιηθεί αυτό το χρηματοδοτικό μέσο και ότι άμεσα πρέπει αυτό το ποσό να διατεθεί στους Ισπανούς εργαζόμενους. Το πακέτο μέτρων είναι 1.400.000 ευρώ, από τα οποία η Ένωση μέσω αυτού του Ταμείου Προσαρμογής για την Παγκοσμιοποίηση θα συνεισφέρει 50%, 700.000 ευρώ. Πράγμα το οποίο θα βοηθήσει τους πάνω από 500 αυτούς εργαζόμενους για να βρουν μια νέα θέση απασχόλησης με μια σειρά υποστηρικτικών μέτρων που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Αυτοί οι εργαζόμενοι υπέστησαν πλήγματα από τα μεγάλα τις μεγάλες διαθροτικές αλλαγές στο διεθνέ εμπόριο που προκραλούνται και προκλήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση και επιπλέον και από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση που είχε όπω γνωρίζετε πολύ αρνητικέ επιπτώσει για την απασχόληση στο σύνολο τη Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ισπανία. Όπω μπορείτε να δείτε στην έκθεση που σα υποβάλλω ο όγκο εξαγωγών από πλευρά ξύλου και φελού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με τα πιο έντονα έτη της ε, κρίσης 2010-2011. Σε αυτή την περίοδο η μείωση στην Ισπανία ήταν ακόμα μεγαλύτερη μια και είχαμε τριπλάσιο αριθμό ε, των ε, επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στην Καστήλη η απώλεια απασχόλησης από το κλείσιμο αυτών των τριών επιχειρήσεων του τομέα ξύλου που έχει επίπτωση σε 587 εργαζόμενους έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην εργασιακή αγορά την τοπική. Ως μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Προϋπολογισμού και ως Ισπανός είναι θεμελιώδες νομίζω να δώσουμε μια άμεση απάντηση και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτούς τους εργαζομένους εργαζομένους. Μια και προέρχονται από μια περιοχή όπου η κατάσταση από πλευράς εργασίας είναι ιδιαίτερα ευάλωτη και είναι μια ζώνη που συνδέεται έντονα με τον τομέα του ξύλου παραδοσιακά και με ένα χαμηλό αριθμό όσον αφορά τον ε, αριθμό κατοίκων και το κλείσιμο επιχειρήσεων οδηγεί σε αποψήλωση πληθυσμού που οδηγεί και σε ε, επιδίνωση των προοπτικών. Γι' αυτό ολοκληρώνω λέγοντας πρόεδρε όλοι αυτοί οι όροι και δεδομένου το ότι υλοποιεί τους όρους η Ισπανία για να τύχει της βοήθειας ε, του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θεωρώ ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει άμεσα να εγκρίνουν την κινητοποίηση αυτών των 700.000 ευρώ που είναι το 50% του συνολικού προϋπολογισμού που θα στοχεύει στο να υλοποιηθούν μέτρα ένταξης στην αγορά εργασίας αυτών των ε, εργαζομένων. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω χωρίς να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις βελτιώσεις που επετέφθησαν στη διαδικασία λήψης απόφασης. Εμένοντας ε, στο ότι αυτή η διαδικασία ε, και ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα εξέχοντα μέλη αυτής της κοινοβουλευτικής επιτροπής ε, και από διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες πέτυχαν αυτό το αποτέλεσμα. Οι Ισπανοί εργαζόμενοι χρειάζονται άμεσα αυτές τις βοήθειες για να μπορέσουν να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Γι' αυτό ζητώ αυτή την υποστήριξη. Πρέπει να πάψει πια να υπάρχει υπάρχει αυτή η μάστιγα της ανεργίας ε, που πλήττει τους εργαζόμενους. Ε, ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση όταν είναι εργαζόμενοι μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και περιοχών που λόγω έλλειψης πληθυσμού, μειωμένου πληθυσμού έχουν πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες για να διασφαλίσουν το μέλλον τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur le rapporteur. Merci. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία παρουσιάσατε και για την πυθό με την οποία παρουσιάσετε τα ζητήματα αυτά. Την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή μας θα χρειαστεί να ψηφίσει για την έκθεσή σας. Θα συνεδριάσουμε την 5η 11 Σεπτεμβρίου και με την ευκαιρία αυτή θα ψηφίσουμε και για την έκθεσή σας λοιπόν. Στη συνέχεια, κατά την Ολομέλεια, θα υποβληθεί η έκθεση αυτή στις 18 Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα. Υπάρχουν ερωτήσεις, παρατηρήσεις προς τον εισηγητή. Όχι. Επομένως μπορούμε να περάσουμε... Συγγνώμη, δεν σας είδα. Ε, Έχετε το λόγο. Only actually one question, Μία ερώτηση μόνο έχω. Είναι διαδικαστικής φύσης. και αφορά όλα αυτά τα αιτήματα. Αν έχουμε ένα αίτημα, για παράδειγμα, από την Φιλανδία, θα μπορούσα εγώ να γίνω εισηγήτρια για το αίτημα αυτό. Διότι εφόσον αφορά τη Φιλανδία, με αφορά το ζήτημα αυτό, θα ήθελα να μπορούσα να εξασφαλίσω και για τη χώρα μου τα χρήματα αυτά. Προβλέπετε λοιπόν μια τέτοια διαδικασία, θα μπορούσα εγώ να λάβω ένα τέτοιο αίτημα. Πρόεδρος, κοιτάξτε, από διοντολογικής πλευράς καταρχάς πρέπει να εξετάσουμε την έκθεση αυτή εντελώς αυτόνομα και ανεξάρτητα και να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τις βασικές αρχές με τρόπο ισότιμο. Ξέρετε ότι προέρχεστε από τη χώρα αυτή, θεωρείτε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει τελικά την εξαρτησία με την οποία αξιολογείται το ζήτημα. Ο κύριος Φερνάντες έχει το λόγο. Δεν θέλω να ξανανοίξουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα, αλλά θα ήθελα να ενημερώσω την συνάδελφο ότι αυτή η κατάσταση ήδη συζητήθηκε στη συνάντηση συντονιστών και ότι η απόφαση που ελήφθη ήταν σαφής. Και από πλευρά του ΕΛΚ είπαμε ότι υποστηρίζουμε τη θέση. Και τίποτα δεν παρακολεί για έναν, ε, έναν ε, υπήκο μιας χώρας να μπορέσει να συντάξει μια τέτοια έκθεση για θέμα που συνδέεται με την χώρα του. Σε αυτή την περίπτωση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και για το θέμα του προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο ξεχωριστό θέμα για μια χώρα διότι αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητική επίπτωση αν υπάρχει έστω και κάποια μικρή διασύνδεση. Και έτσι δεν πρέπει να υπάρχει κανένα κόλλημα. Το αντίθετο, αξιολογούμε ιδιαίτερα τον ρόλο των Ευρωβουλευτών με αυτόν τον τρόπο. Και αν κάποιος διαφωνήσει από πλευράς αυτού του θέματος μπορεί να υποβάλει τροπολογίες και δεν βλέπω κανένα να έχει αμφισβητήσει οποιοδήποτε θέμα δεοντολογικό ή κάποια έλλειψη δεοντολογική ή ηθική, ηθικού χαρακτήρα για αυτό το θέμα. Το ότι υπάρχουν προηγούμενα δεν είναι το, η πρώτη φορά που γι' αυτό το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση από πλευρά ε, βουλευτού ε, μια αρμόδια χώρα να αναλαμβάνει μια έκθεση έχει ήδη αποσαφινιστεί και ολοκληρωθεί τελεσίδικα αυτό το θέμα μετά από αυτή τη διαβούλευση. Οι ευρωβουλευτές λοιπόν συνήγαγαν τα συμπεράσματά τους ελεύθερα και καταλήγουν σε ελεύθερη δράση. Ως ευρωβουλευτές ε, έχουν ε, σημαντικό ρόλο και είναι σημαντικό να καταδεικνύεται επίσης ε, μέσω του έργου τους ότι υπάρχει αυτή η διασύνδεση ακόμα και με τη χώρα που, για την οποία εκλέγονται. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πλέον σαφές ε, είναι σαφής η θέση μας. Και πιστεύω ότι δεν μπορεί με κανένα τρόπο να προσβληθεί υπονομικού ή ηθικού ή δεντολογικού πρίσματος. Ευχαριστώ. Merci, Monsieur Ο κύριος Ετσενίκου έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ευρώ αν τα μοιράσουμε μεταξύ 400 είναι 10.500 ευρώ ανεργαζόμενο. Και έτσι δεν θα επιληθούν τα προβλήματα της ζωής αυτών των ατόμων που επλήγησαν και έχασαν την εργασία τους εδώ και αρκετούς μήνες ήδη στο παρελθόν. Τούτου λεχθέντος προφανώς πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την κινητοποίηση κονδυλίων άμεσα από αυτό το ταμείο ώστε να ανακουφιστούν. Και έτσι θα υπερψηφίσω σε, όταν θα έρθει η ώρα θα μπορέσω να υπερψηφίσω ως αναπληρωτής. Ωστόσο όμως δεν μπορεί κανείς να το δει διαφορετικά. Πρέπει να λάβουμε την θέση να υιοθετηθεί το πιο αποτελεσματικό μέτρο, ιδιαίτερα για την πρόληψη σε σχέση με την ιατρική ε, οποιονδήποτε ασθενειών. Ίσως θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που απολύθηκαν από τις εργασίες τους ε, να εξετάσουμε σε σχέση με τα εργασιακά όχι μόνο τα εργασιακά, όπως γίνεται σε κράτη-μέλη, αλλά και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαφορετικών θεσμικών οργάνων της να προσπαθήσει να ε, προστατεύσει αυτούς τους εργαζόμενους από τις επιπτώσεις παγκοσμιοποίησης πέρα από την ε, αποζημίωση, αποζημίωση, με ποσά όχι τόσο γενναιόδωρα που δεν μπορούν βέβαια να επιλύσουν τέτοιου είδους προβλήματα όταν έχει ε, ήδη συμβεί μια τέτοια απόλυση που είναι σημαντικό πλήγμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Τον λόγο τον ζήτησα μετά από την παρέμβαση της συναδέλφου μας πιο πριν για το αν είναι επαρκές ή όχι ένας ευρωβουλευτής μιας χώρας να μπορεί να εργάζεται για αυτό το θέμα σε σχέση με το ταμείο αυτό για τη χώρα του. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει και μπορεί κανείς να κάνει ως Ευρωβουλευτής ε, οτιδήποτε επιθυμεί γιατί δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα. Αλλά αν υπάρχει κάποια αμφιβολία <clears throat> οι δυνατότητες που έχουμε ως Ευρωβουλευτές για τι τις δράσεις του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης δεν είναι τεράστιες το να πιστοποιήσουμε ότι υλοποιούνται οι όροι και, οι προϋποθέσεις προς το κράτος από το οποίο προέρχεται το αίτημα αρρωγής. Δεν μπορούμε με άλλο τρόπο εμείς να καθορίσουμε ούτε το ποσό ούτε τι πώς θα γίνει. Είναι λοιπόν σε σχέση με το αίτημα αυτό ελεύθερη η οδός να εργαστεί ένας ευρωβουλευτής ή μια ευρωβουλευτήνα για αυτό το θέμα που αφορά ίσως και την ίδια του τη χώρα και μάλιστα μπορεί να έχει και καλύτερες γνώσεις ε, για τις περιπτώσεις αυτές. Ε, δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να ε, παρακολύσουμε κάποιον, ούτε να ευνοήσουμε κάποιον ο οποίος έχει την πρόθεση να εμπλακεί σε αυτό το θέμα. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με τη δράση για αυτό το ταμείο ή και άλλα ταμεία, παρότι δεν μπορεί να είναι πανάκια για την επίλυση όλων των εργασιακών προβλημάτων στην Ένωση, είναι παρόλα αυτά μια μικρή ανακούφιση, μια μικρή συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθηθούν στην κατάρτισή του, στην εκπαίδευσή τους, στην επιμόρφωσή τους επαγγελματική αυτοί οι εργαζόμενοι που ίσως έτσι θα μπορέσουν να βοηθηθούν, θα μπορέσουν να βοηθηθούν με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Δεπρά έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ δημοσίως να πω τη δική μου την άποψη. Γιατί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών ήμουνα υπέρ της άποψης που ανέφερε αυτή τη στιγμή η κυρία Μακή. Αλλά πρέπει να σας πω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί συντονιστές οι οποίοι τάχθηκαν υπέρ της άποψης που πρεσβεύει αυτή τη στιγμή η συγγήτρια, η γενική μας μάλλον συγγήτρια για τον προπολογισμό. Ενδεχομένως ε, να μην ε, είχε ενημερωθεί η ε, συνάδελφος η οποία πήρε το λόγο πριν από λίγο. Δεν είχε ενημερωθεί ουσιαστικά για τόσα υπόθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας των ιστών. Αν λαμβάνουν λοιπόν την ευθύνη. Ο κύριος Κολβέλ έχει το λόγο. Ναι, μόνο σύντομα θα προσθέσω κάτι αν επιτρέπετε, επειδή έχω την εντύπωση ότι κάποιες παρεμβάσεις που έγιναν νομίζω υπερβολικά στοχεύουν προς το θέμα ουσίας Είμαστε εδώ Επιτροπή Προπολογισμών και από ό,τι γνωρίζω στην Επιτροπή Προπολογισμών συχνά πρέπει φρικτά πράγματα από πλευρά δημοσιονομική εμεί να υιοθετούμε. Ωραίο θα ήταν να μπορούσαμε όλα τα προβλήματα να τα επιλύαμε με χρήματα, αλλά δεν έχουμε ούτε τόσο μεγάλα ποσά, ούτε μπορούμε να είμαστε πιο γενναιόδοροι στο μέλλον. Θα ήταν εξάλλου και σφαλμένο μήνυμα, λαθασμένο μήνυμα από την Επιτροπή Προπολογισμών. Κάτι τέτοιο να περνούσαμε προ τα έξω, ότι αυτή είναι η δουλειά μα. Ότι και αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, πάντα αρκετά κονδύλια θα μπορούσαν να διατεθούν από πλευράς μας. Διότι το θεωρώ περισσότερο ως ένα ταμείο πυροσβεστικό, ώστε οι πιο έντονες ανάγκες να μπορέσουν να ανακουφιστούν από, μια τέτοια, από τέτοια πλήγματα. Αυτό είναι απλώς μια, όχι θεραπεία, αλλά μια αντιμετώπιση συμπτωμάτων μόνο. Γι' αυτό έτσι πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Ο κύριος εισηγητής και πάλι. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για την υποστήριξη των όσων παρενέβησαν σε αυτή τη συζήτηση για την απελευθέρωση των κονδυλίων αυτής της βοήθειας αρρωγής προς την Ισπανία. Να πω δύο πράγματα για να ολοκληρώσω. Πρώτα απ' όλα, για να αποσαφηνίσω ένα αμφίσιμο θέμα από τον συνάδελφο από την αριστερά. Είναι ένα ταμείο που θέλει να επανακαταρτήσει και να βοηθήσει στην επανακατάρτιση ατόμων που έχασαν την απασχόλησή τους. Όχι να τους αποζημιώσει για να μπορέσουν λοιπόν να επανακαταρτιστούν, να επιμορφωθούν για να μπορέσουν να βρουν μια νέα ε, ε, εργασία. Πρέπει να γίνει κατανοητό ποια είναι η φύση του θέματος που συζητούμε, ώστε οι αντιδράσεις μας να μπορούν να στοχεύουν προς τον ορθό ε, τομέα. Για την συνάδελφο από την Φινλανδία, δεν είναι ελάσσονο σημασία στο θέμα που θίξατε. Αφορά την ίδια την ουσία της εργασίας μας εδώ στην Ευρωβουλή. Δεν είμαστε εμείς κριτές ή δικαστές. Δεν είμαστε εμείς η διοίκηση. Είμαστε συνήγοροι των πολιτών μας. Είμαστε ευρωβουλευτές και προασπίζουμε και εκφράζουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας. Εγώ υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των δικών μου ψηφοφόρων Είμαι βέβαιος ότι αν ήταν θέμα για την Φινλανδία, εσείς θα υποστηρίζατε τα θέματα των Φινλανδών. Και δεν είναι ένας ευρωβουλευτής που λαμβάνει τις αποφάσεις, είναι όλοι μας, εσείς και εμείς. Αυτό που προτείνει ένας εισηγητής ψηφίζεται, τίθεται υποψήφιση σε μια ε, κοινοβουλευτική επιτροπή. Δεν είναι ατομική απόφαση ενός ευρωβουλευτή. Αυτό που κάνει ο ευρωβουλευτής είναι να έχει την τιμή να υπερασπίζεται τους ψηφοφόρους του. Αυτό έκανα και εγώ εδώ ως εισηγητής. Ευχαριστώ. Eh Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιείται μόνο όταν τελικά αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις όπου έχουν ε, μετεγκατασταθεί δραστηριότητες μιας επιχείρησης, αν θέλουμε να αποφύγουμε το φαινόμενο αυτό, τότε νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλους διαφορετικούς τρόπους για να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα σε μια περιοχή και να αποφύγουμε όλες αυτές τις πολλές δεινές κοινωνικές συνέπειες. Όπως είπε ο κύριος Κόλμερ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμοποίηση χρησιμοποιείται ως ε, ίστατη λύση τελικά, ως έσχατη λύση, μόνο όταν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τίποτα άλλο. Στις 11 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί λοιπόν η σχετική ψηφοφορία και θεωρώ ότι ε, ο εισηγητής κατάφερε να μας διαφωτίσει σε σχέση με την απόφαση που θα πάρουμε λοιπόν στις 11 Σεπτεμβρίου. Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης. Δίνω το λόγο στον κύριο Νίλς Τόρβατς, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του, το οποίο υπευλήθη στις 29 Αυγούστου στα μέλη της Επιτροπής μας και ουσιαστικά συνεχίζει την ε, σειρά αυτή των γνωμοδοτήσεων που έχει υποβάλει η Επιτροπή Προπολογισμών όσον αφορά το ζήτημα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και αυτή τη φορά αναφερόμαστε βέβαια στο 2014. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη φορά θα είμαι αρκετά σύντομος. Ε, δεν μιλάμε για την ε, υλοποίηση των προτεραιοτήτων του προπολογισμού του 2014 έχει σχέση με την έκθεση της ΕΚΟΝ επί του δύο θέματος και ελπίζω ότι θα διαβάσετε και τις δύο εκθέσεις για να πάρετε τη σωστή προσέγγιση. Η, γνωμοδότηση επισημαίνει την σημαντική, το σημαντικό ρόλο του ευρωπαϊκού προπολογισμού για την υποκίνηση της ανάπτυξης. Υπενθυμίζει ότι η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών ε, μπορεί να ε, ε, χρησιμοποιήσει το σύστημα ιδίων πόρων που μπορεί να περιορίσει τα προβλήματα. Ξέρετε την, όλη την Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου προσπαθεί να δώσει λύση αυτό το πρόβλημα πρόβλημα, όλοι περιμένουμε κάτι από αυτή την πηγή. Και όσον αφορά την ε, συζήτηση για το προπολογισμό του 2015, ήδη από ε, σήμερα το πρωί υπάρχουν ε, ενισχυτικές ενδείξεις και για το ξεκίνημα νέων προγραμμάτων και από την Επιτροπή ΠΑΣΚ. Επίσης στην έκθεση Baker υπάρχουν θέματα που μας αφορούν και εδώ. Αλλά επειδή ε, και οι δύο αναφέρονται θα παρακαλώ να ληφθούν υπόψη. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 15η Σεπτεμβρίου και ελπίζουμε ότι στις 30 θα μπορέσει να ψηφιστεί η γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ πολύ ε, για την ανακοίνωση αυτή. Υπάρχει, υπάρχουν παρατηρήσεις ο κύριος Φερνάντες. Πολύ σύντομα. Εξ ονόματος της συναδέλφου Γκράσλερ που δεν μπορεί να είναι παρούσα για να συγχαρεί να συγχαρούμε τον εισηγητή κύριο Τόρβατς για αυτή την έκθεση που έχει υποβάλει, τη γνωμοδότησή του. Και υπάρχει συμφωνία γενικότερη για τις προτάσεις που διατυπώνει και τα θέματα που ανέφερε επί των οποίων τοποθετήθηκε. Ο προϋπολογισμός πρέπει να δίνει κίνητρα για την ανάπτυξη, είναι προφανές αυτό και για την ανάγκη να κινητοποιηθούν αυτό το έτος και να λειτουργήσουν τα πολιτή δημοσιονομικά πλαίσια MFF για να προαχθεί η απασχόληση, ιδιαίτερα η απασχόληση των νέων να δράσουμε ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την ενεργειακή μας εξάρτηση και τα διαθωτικά ταμεία και κονδύλια στο επίπεδο των κρατών μελών να μπορέσουν να οδηγήσουν σε μεταρρυθμίσεις διαρθρωτικές σε όλη τη ζώνη ευρώ συνολικά. Υπάρχει μεγάλη διασύνδεση και αλληλεξάρτηση όπως έχει επανειλημμένα ε, καταδειχθεί για να προαχθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις και να υπάρξει η ανάπτυξη όπως η συνάδελφος Γκρέσλερ θα ήθελε και εκείνη να προτείνει και να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν τα ίδια με καλύτερο τρόπο την χρήση των κονδυλίων για την ανάπτυξη, για την απασχόληση και για την αύξηση, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Είναι προφανές ότι αυτό το αίτημα επίσης το συνειδητοποιούμε και υπάρχει ανάγκη τα θεσμικά όργανα να δράσουν και να υλοποιήσουν. Και αυτά τα οποία συζητώνται εδώ σήμερα επίσης και για την κάλυψη των ε, πιστώσεων πληρωμών, την υλοποίηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουμε για την επίτευξη αυτού του σκέλους των υποχρεώσεών μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία που έχει επιτελέσει για τη γνωμοδότηση αυτή, με την οποία ουσιαστικά συμφωνώ. Και εγώ όμως θα ήθελα αυτή τη στιγμή να καταθέσω κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, βλέπουμε ότι έχουν περάσει εδώ πάρα πολλά χρόνια πλέον όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέει ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο κοινοτικό προπολογισμό προκειμένου να καταφέρουμε να υποστηρίξουμε την οικονομία και την απασχόληση στα κράτη-μέλη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε όμω ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη υπονομεύουν τελικά το κοινοτικό προπολογισμό κάνοντα συνεχώ οριζόντιε περικοπέ. Συμφωνώ λοιπόν με τι προτάσει που γίνονται εδώ πέρα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβουμε στην ετήσια επισκόπηση τη ανάπτυξη ακόμα και τι επιπτώσει που έχει ο κοινοτικό προπολογισμό όσον αφορά τι εθνικέ δημόσιε δαπάνε. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθούμε και στι τοπικέ και περιφερειακέ δαπάνε είναι πολύ σημαντικό κάποιε πρωτοβουλίε όπω η εγγύηση για την νεολαία να μην θεωρούνται ότι αποτελούν επιβάρυνση για τι δημόσιε δαπάνε. Προφανώ θέλουμε τα οικονομικά μα να είναι υγιή. Προφανώ θέλουμε να έχουμε Ευρωπαίου πολίτε οι οποίοι παράγουν και εργάζονται. Προφανώ θέλουμε νέου οι οποίοι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν τελικά τι ιδέε του και να πραγματοποιήσουν το ταλέντο του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία μα. Και για άλλη μια φορά θα ήθελα να σα πω το ακόλουθο. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν τελικά να μειώσουν τι συνεισφορά του στον εκνοτικό προπολογισμό έτσι ώστε τελικά να διευκολύνεται περισσότερο ο έλεγχος των δαπανών, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο σύστημα ή θα μπορούσε μάλλον να διευθετηθεί αυτό με ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων. Πάρα πολύ συχνά το έχει ζητήσει αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητάμε λοιπόν από την ομάδα εργασία Μόντι πλέον μια φιλόδοξη, πιο θαραλέα πρόταση, η οποία πραγματικά να καταρτήσει ένα νέο σύστημα ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι με τι αποφάσει που ελήφθησαν το τελευταίο διάστημα δεν έχει βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Χάνονται συνεχώ θέσει απασχόληση. Όλο και περισσότερε είναι επιχειρήσει οι οποίε κλείνουν. και αυτό έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει για την σταθερότητα. Είναι σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε κάποιε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει, αλλά παράλληλα επίση και κάποιε σημαντικέ επενδύσει προκειμένου να οδηγηθούμε σε οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Χωρί τι επενδύσει αυτέ δεν θα καταφέρουμε να φτάσουμε ποτέ στο επίπεδο ανταγωνιστικότητα των άλλων κρατών εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλε αυτέ οι πτυχέ, όλη αυτή η διάσταση να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α μην ξεχνάμε ότι ο κοινοτικό προπολογισμό έχει έναν πολύ ευνοϊκό ρόλο για την ανάπτυξη της οικονομίας των κρατών μελών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν όλες οι χώρες και οι χώρες Ευρωζώνης να προχωρήσουν στις κατάλληλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ανάπτυξη και ουσιαστικά θα αποφύγουμε κατά αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουμε ένα τεράστιο χρέος το οποίο θα βαρύνει τις επόμενες γενναίες. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κάποιο άλλο το λόγο. Οπότε... Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τροπολογίες για την ε, έκθεση αυτή πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα και ότι η Επιτροπή ε, θα ψηφίσει κατά συνεδρίαση της 30 Σεπτεμβρίου. Στο σημείο αυτό Εξαντλήσαμε την ημερική διάταξη. Οπότε στρέφομαι σε εσά. Αν υπάρχουν διάφορα. Υπάρχει κάποιος που ζητά το λόγο για τα διάφορα. Μοιάζει πως όχι. Φυσικά θέλω να παραμείνουν οι συντονιστές γιατί σήμερα το πρωί διακόψαμε για να γίνει η συνεδρία της Επιτροπής. Οπότε σας ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας στα δύο αυτά τμήματα της συνεδρίας της, Επιτροπής Επόμενη συνεδρίαση την 5η 11 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί εδώ στις Βρυξέλλες. Λύεται η συνεδρίαση για όλα τα μέλη της Επιτροπής με εξαίρεση τους συντονιστές.